είναι ο κύριος Κλοντ Ρολάν. Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία που αφορά την απόσπαση εργαζομένων είναι ένα θέμα εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο για τους εργαζόμενους αλλά και για τους ε, διευθυντές επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών και των οδικών μεταφορών. Ε, καθημερινά έρχονται σε επαφή μαζί μου πολίτες αλλά και εργοδότες. Ε, το κοινωνικό dumping είναι μια, ένα πραγματικό, μια πραγματική πληγή που αναπτύσσεται η απόρριψη ε, του ευρωπαϊκού οράματος. Πρέπει πραγματικά να καταπολεμηθεί και σταθερά να καταπολεμηθεί. Η οδηγία αυτή διορθώνει κάποιες αδυναμίες αλλά πρέπει επιγόντως να μεταγραφεί στις εθνικές νομοθεσίες και αυτό μάλιστα με φιλόδοξο τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των μισθωτών και να τεθεί ένα τέλος στις καταχρήσεις και στην, ε, στον αθέμετο ανταγωνισμό. Ε, οι ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να βασιστούν στην πείρα και στη γνώση των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει μέσα να σκεφτούμε τον τρόπο μερικής αναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τσάμπα Μόλναρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Χωρίς μικρόφωνο μιλητή. Εντάξει, τώρα δουλεύει. Ναι, ναι, μπορείτε να μιλήσετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με το εξή. Δεν θέλουμε ανθρώπους με διαφορετικούς ε, πολιτισμούς ε, γύρω μας. Θέλουμε η Ουγγαρία να μείνει Ουγγαρία. Αυτό δεν το είπε κάποιος ακραίος, ε, αλλά ο Πρωθυπουργός μας, ο Βίκτορ Όρμπαν, στο Παρίσι χτες. Πρόκειται για κάτι το φρικτό και ρατσιστικό. Προσβάλλει τους Γάλλους και την μνήμη των νεκρών. Ο Πρωθυπουργός μας θεωρεί τους μετανάστες την ρίζα κάθε κακού, απέδειξε και πάλι πως δεν έχει θέση μεταξύ των άλλων ηγετών. Ήμουν στο Παρίσι και στόχο δεν είχε να αποκλείσει κάποιον. Ε, στόχος ήταν να υπερασπίσει τις αξίες και τις ιδέες. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν μίλησε εξ ονόματος όλων των Ούγκρων. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Άγχελ Τσαμπάσκι για ένα λεπτό επίσης. Κύριε Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το... Τα πρόσφατα γεγονότα στο, Παρίσι, στο Παρίσι, τρομοκρατική, ισλαμιστική επίθεση ε, κατά των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με κάνει ανησυχώ για τις προοπτικές ε, χιλιάδων ε, παράνομων μεταναστών που μπαίνουν στην Ευρώπη και από τη Βουλγαρία μάλιστα. Τα πρόσφατα γεγονότα απαιτούν να ξανασκεφτούμε το σύστημα ε, μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και των κοινών μας αξιών. Η Βουλγαρία δεν μπορεί να συντηρεί στο εδάφιο της ε, χιλιάδες παράνομους μετανάστες που δεν έχουν λάβει το καθεστώς πρόσφυγα. Χρειαζόμαστε πολιτική, κοινή πολιτική μάλιστα ασφάλειας και μία ε, ρύθμιση που θα μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλειά μας και την ασφάλεια των αξιών μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεσέρα Μπαστερέτσια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στη Βενεζουέλα υπάρχουν πολιτικέ διώξει, λογοκρισία των ε, μέσων, ε, παράνομε φυλακίσει, ε, βασανισμοί και δολοφονίες των μελών τη αντιπολίτευση. Αυτή δεν είναι μια γνώμη, είναι η πραγματικότητα. Ε, χώρες ε, ε, όπως το Βέλγιο αναγνώρισαν αυτές τις πολιτικές ε, διώξεις. Ο Λεοπόλδο Λόθεθ παραμένει φυλακισμένος. Το Κοινοβούλιο καταδικάζει κατ' επανάληψη αυτή την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι ευρωβουλευτές αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν το ψήφισμα θα πρέπει ωστόσο ε, να γίνει αυτό το βήμα ούτως ώστε η κυβέρνηση της ε, Βενεζουέλας να αναλάβει τις ευθύνες της και να δρώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, υπάρχουν πολλοί πολίτες θα αντισταθούμε σε αυτή την ε, κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Νεοκλής Ηλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις 6 Ιανουαρίου η Τουρκία συνεχίζοντας τις παράνομες ενέργειες έκδοσε νέα οδηγία Ναύτεξ προς ναυτιλιωμένους με την οποία δεσμεύει περιοχές στην ανατολική μεσόγειο εντός της Κυπριακής αποκλειστική Οικονομικής Ζώνης για να διεξάγει έρευνε μέχρι τις 6 Απριλίου. Η ελέγχο ενέργεια τη Τουρκία καταπατεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπονομεύει τις προσπάθειες για επανέναρξη της διαδικασία για του Κυπριακού. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δρανεί, πρέπει να αξιοποιηθεί το πρόσφατο ψήφισμα της Ευρωβουλή, για το οποίο καλείται η Άγκυρα να αποσύρει την παράνομη οδηγία και να απομακρύνει το ερευνητικό πλοίο τη και τη συνοδεία από την κυπριακή αός. η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να πιέσει την τουρκία να πάψει να παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών αλλά και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιριών eni και total οι οποίε διεξάγουν ερευνητικέ γεωτρήσεις εντό τη κυπριακή αός. αναμένουμε από την ευρωπαϊκή ένωση να πάρει άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα ώστε η τουρκία να αποσύρει την ναύτεξ και να σταματήσει οποιαδήποτε προκλητική και παράνομη ενέργεια. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χόρντι Σεμπαστιά. Κυρίες κολέγας, Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 15 Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία έκανε, έφερε ένα καλό νέο για τους ασθενείς ε, της ε, υπατήτηδας ΣΕ. Υπάρχουν νέα σκευάσματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Ωστόσο, η χαρά, τη χαρά αυτή δεν μπορούν να τη συμμεριστούν οι πολίτες της Ισπανίας, γιατί η κυβέρνηση ε, περιόρισε την ε, χρήση αυτών των φαρμάκων ε, σε μια μικρή, σε ασθενείς, παρόλο που καθημερινά πεθαίνουν ασθενείς στην Ισπανία που πάσχουν από υπατήτηδα γάμα. Ε, και αυτό έγινε λόγω της ε, πίεσης των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών που βάζουν το κέρδος πάνω από το όφελος της υγείας των Ισπανών ε, πολιτών. Και εάν πραγματικά η Ευρώπη επιτρέψει οι πολίτες της να πεθάνουν λόγω των συμφερών των μεγάλων εταιριών θα γίνει συνένοχός τους. Λένε πως πρέπει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ε, θέσεις εργασίας. Αυτά πείτε τα 220 ψηφοφόρους μου που έχασαν τη δουλειά τους όταν έκλεισε το 2013 ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτά χάρη στην οδηγία σας ε, που κλείνει η εργοστάσια που μας δίνει το 1 τρίτο της ενέργειάς μας. Ε, τα πυρηνικά εργοστάσια ενώ ο Ed Miliband ήταν υπουργό Ενέργειας. Μου ζήτησαν οι ψηφοφόροι μου λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Μίλιμπαντ και τους υπόλοιπους γιατί δεν έκαναν τίποτα για τις δουλειές αυτές. Μας κοστίσατε θέσεις εργασίας. Οι μέρες που το εργατικό κόμμα φρόντιζε τους εργαζόμενους έχουν παρέλθει. Έχετε ξεχάσει κοινότητες όπως το Τίλμπερι και το Θάροκ και τον Μάιο θα σας κρίνουν με βάση τις πράξη σας, γιατί πλέον δεν εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ. Σόλταν Μπάλτσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το θα ο South Stream, South προσφέρει μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη. Όμως ε, οι κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν να γίνει αυτός ο αγωγός. Όμως ε, το να πηγαίνει αέριο στη Γερμανία μόνο δεν αποτελεί πρόβλημα. Επιτετραμένος ε, τον είπα στην Ουγγαρία λέει πως το streamline ε, της Ουγγαρίας, το αγωγός αυτός ε, απειρεί απειλεί τα συμφέροντά τους. Πρέπει να αποφασίσουν επιτέλους ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή πιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Όταν μιλάμε για παγκόσμιο ανταγωνισμό συμφερόντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ ή, ή κάποιο άλλο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαριάννα Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή λιπολής λόγος γίνεται για το κράτος δικαίου, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από Σερβία να αλλάξει την ομοθεσία της για την σύσταση κρατικών οργάνων στις δίκες περί εγκλημάτων πολέμου. Αν δεν γίνει αυτό δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί απειλούνται τα συμφέροντα Κροατών πολιτών. Η Σερβία προσπαθεί και δικάζει ε, Κροάτι πολίτη για έγκλημα που έγινε εναντίον άλλου Κροάτι πολίτη σε κροατικό έδαφος. Πράγματα παράλογα δηλαδή. Ο Βέλικο Κροάτης ε, στρατιώτης απήχθη στην Σερβία, τον ε, κρατούσαν επί πέντε χρόνια εκεί πέρα και απαιτώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τη Σερβία να καταργήσει αυτόν τον ε, νόμο και ο κύριος Μάριτς να μεταφερθεί στην Κροατία και να έχει μια δίκαιη δίκη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιέζη Πόσπισιλ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους πως έχουμε ένα νέο νόμο στη χώρα μου πήγε περί δημοσίων προμηθειών ο οποίος ε, νομίζω ότι παραβιάζει την σχετική κοινοτική οδηγία του 2014. Προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ειδικά στα θέματα των δημοσίων προμηθειών και να στηρίξουμε επιχειρηματίες οι, οποίες, οι οποίοι θέλουν να αναζητήσουν εργασία και να αναλάβουν έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στην ε, χώρα τους. Αν προσεγγίσουν λοιπόν οι κανόνες αυτοί θεωρώ πως ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερες δυνατότητες για να εργαστούν πανευρωπαϊκά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την οδηγία και θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά το δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών. Ευχαριστώ. Η κυρία Κατρίν Στήλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα σήμερα να μιλήσω για το φρικτό έγκλημα της, του δουλεμπορίου και της, του εμπορίου παιδιών. Το δουλεμπόριο είναι η πιο γρήγορα αυξανόμενη οικονομία στον κόσμο. 1,2 εκατομμύρια κόσμους ε, διακινούνται παγκοσμίω και εκτιμάται ότι μεταξύ των 27 και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι, είναι παγιδευμένοι σε μια ζωή δουλείας. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την εκστρατεία No Child Taken που ακριβώς εστιάζει σε αυτό το θέμα και στα δικαιώματα των πιο ευάλωτων παιδιών, τη βοήθεια προς αυτά ε, με παιδεία, ε, κατάρτιση για να μπορέσουν αυτά ε, να ελπίζουμε ότι αυτά τα παιδιά θα γλιτώσουν από το δουλεμπόριο. Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πέφτει θύμα εμπορίου και την ώρα που μίλησα τρία παιδιά ήδη έχουν ε, πέσει θύματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναχαιτήσουμε αυτά τα φρικτά εγκλήματα και να εξασφαλίσουμε την προστασία των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, κυρία Στήλερ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Άλφρετ Σαντ. Σας ευχαριστώ τα πρόσφατα χρόνια έχουμε φτιάξει έναν ε, χώρο ασφάλειας για το ευρώ. Καλύτερα ε, όργανα μέσα για να μπορούμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά μας ε, αποτελέσματα. Αυτό έδωσε την εντύπωση πως τα πράγματα είναι υποέλεγχο. Γιατί λοιπόν τότε οι εξελίξεις που υποτίθεται είναι σχετικά μικρής ε, σημασίας όπως οι εκλογές στην Ελλάδα έχουν, δημιουργούν τόσες πολλές ανησυχίες. Η Ευρωζώνη έχει γίνει πολύ σπουδαία, too big to fail, πολύ μεγάλη για να αποτύχει. Ε, το, το σχέδιο αυτό έχει οικοδομηθεί επί τη βάση του soft power της οποίας χαίρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχει τις κατάλληλες ομοσπονδιακές στο δομές ώστε το ευρώ να είναι ε, σταθερό και συμπαγές. Εν τω μεταξύ, η χρήση τεχνικού θετικισμού για τον έλεγχο της κατάστασης μετατρέπεται σε μια άσκηση πολιτικού φετιχισμού που μπορεί να υποβαθμίσει την ε, δύναμη και την ισχύ της, της Ένωσης. Σε πολλές ε, από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωζώνης βασίζονται σε ξεπερασμένες θεωρίες. Πρέπει να ανανεωθούν. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ιωάχιμ Σταρμπάτη. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι που έζησα στο γραφείο μου στις ε, Βρυξέλλες, κάτι που συμμερίζονται κατά πάσα πιθανότητα πολλοί από εσά. Ε, ε, ενώ βρίσκομαι στον υπολογιστή μου, κόβεται το ρεύμα ε, πάω στο διακόπτη και σκοντάφτω στο καλώδιο. Ε, μαγικά, όχι μαγεία, ανάβει το φως και αυτό επαναλαμβάνεται. Ε, τι γίνεται. Στο γραφείο μου υπάρχει ε, μια συσκευή η οποία ελέγχει κατά πόσο το ρεύμα ε, θα πρέπει να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Δεν νομίζω αν ε, με τον τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματική εξοικονόμηση. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι το ευκταίο να κουνάμε τα χέρια μας ε, στο γραφείο των ε, Βρυξελών για να δείξουμε ότι είναι παρόντες. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αθλητικές ε, ασκήσεις το βράδυ στα γραφεία μας στις Βρυξέλλες για να εξοικονομείται ρεύμα θα το ελέγξουμε. Ένας άλλος τρόπος να αφλείται κανείς είναι να πηγαίνει, να μεταβαίνει από ένα γραφείο των Βρυξελών στο άλλο. Και αυτό είναι ένα ωραίο σπορ, απαντάει η Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής... Η ε, τα γεγονότα είναι, είναι αυτά που υπήρξαν και βρίσκομαι κάτω από το μεγάλο σοκ της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι. Μία τρομοκρατική επίθεση η οποία καταδικάστηκε από τον πρόεδρο του Φιλεύθερου Κόμματος ε, λέγοντας ότι ε, ότι είναι η πολυμορφία αυτή η οποία θα πρέπει να αποτελέσει μια απάντηση στην ε, τρομοκρατία. Θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο ε, είχε συμβεί στην ε, Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της συνόδου της, του Νοεμβρίου. Μια διαπίστωση που έκανε η εκλογική επιτροπή στη χώρα μου επειδή εγώ ε, χρησιμοποίησα κάποιες λέξεις από τη μητρική μου γλώσσα μαζί με τα βουλγαρικά. Ε, κατ' ουσία αυτό αποτέλεσε μία παραβίαση του άρθρου 9 για την ε, προστασία των εθνωτικών μειονοτήτων και των άρθρων 11 και 12 την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και πραγματικά αναφέρω αυτό το συμβάν γιατί επιθυμώ και η χώρα μου να βρίσκεται στο ύψος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Σματ Κάρθη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για να εξαναγκαστούν οι Ιρλανδοί να πληρώσουν ε, το 43% της ε, κρίσης οι τράπεζες έχουν ε, επιβάλει πάρα πολλές κρυφές χρεώσεις και φόρους. Ε, όλα αυτά δεν οδήγησαν σε καλύτερες υπηρεσίες, ήταν απλά άδικες ε, χρεώσεις και, φόρους, και φόροι και βεβαίως πλήττουν δυσανάλογα αυτούς με χαμηλά εισοδήματα. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, κατέβηκαν σε πορεία κατά του τελευταίου φόρου, το οποίο λέγεται τέλος νερού. Αλλά οι Ιρλανδοί ξέρουν τι είναι. Άλλος ένας φόρος που πλέον αν επιβληθεί θα οδηγήσει πάρα πολλές οικογένειες ε, στα όρια τους. Τώρα όμως ε, υπάρχουν και προσωρινά ε, πλαφών. Κάτι το οποίο αποδεικνύει πως ε, δεν υπάρχει σχέση με το να γίνει εξοικονόμηση νερού. Θα πέσει αυτός ο φόρος υδάτων και θα, γίνει, θα δημιουργηθεί μια νέα Ιρλανδία που θα έχει ξεπεράσει αυτή την ατζέντα της λιτότητας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καρίμα Δελή. Chers collègues, hier Αγαπητοί συνάδελφοι, χτε στο Παρίσι και σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο ήμασταν εκατομμύρια που είπαμε δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ υπερασπιζόμενοι τις αξίες μας, κατά των επιθέσεων, ε, κατά της ελευθερίας έκφρασης, ε, κατά ε, της δυνατότητες να συμβιώσουμε. Εμείς θέλουμε να συμβιώσουμε και αυτή η βούληση είναι μια ευκαιρία. Μετά από το φόβο που περάσαμε χθε ζήσαμε την ενότητα μέσα στην διαφορά και δείξαμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί αυτή την περιπέτεια. Περισσότερο από ποτέ ας φτιάξουμε μαζί την Ευρώπη, μια Ευρώπη για όλους, μια Ευρώπη όπου ο καθένας και καθεμιά θα έχει το χώρο του της, ε, όπου κανένας δεν θα αισθάνεται ότι απειλείται επειδή είναι δημοσιογράφος ή επειδή είναι Εβραίος ή επειδή είναι ε, μουσουλμάνος, επειδή είναι αστυνομικός ή μετανάστης. Ορισμένοι φοβούνται τις γενικεύσεις, άρα φοβούνται για την ασφάλειά τους, αλλά αυτός ο φόβος είναι κατανοητός δεδομένων των γεγονότων των τελευταίων ημερών. Αλλά πρέπει να τους πούμε δυνατά και ε, μεγαλόφωνα ότι δεν φοβόμαστε, είμαστε όλοι μαζί, δεν φοβόμαστε να οικοδομήσουμε το μέλλον της κοινωνίας μας και θα το πω και στο τέλος μια μεξικανική παροιμία. Θέλησαν να μας θάψουν αλλά δεν κατάλαβαν ότι ήμασταν σπόροι, σπόροι δημοκρατίας και ελευθερίας. Σας αναλάβουμε λοιπόν τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αντελή. Η κυρία Τζούλια Μόη είναι επόμενη μιλήτρια. Αξιότιμη Πρόεδρε, εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σε τον κίνδυνο που πλήττει ένα μικρό νησί στο κέντρο της Μεσογείου που είναι γεμάτο από σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, στη Σαρδινία. Η Σαρδινία μπορεί να καλυφθεί από ραδιενεργά απόβλητα. Αφού έβαλαν ε, εκεί στρατικές βάσεις ε, όπου χρησιμοποιήθηκαν και αποθηκεύθηκαν πυρηνικά όπλα, ε, τώρα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των πολιτών και και ε, πυρνικά απόβλητα. Η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει πώς και πού ε, έχουν αποθηκευθεί τέτοια απόβλητα. Θα πρέπει η Ευρώπη πρώτη να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποφύγει αυτό το φρικτό ε, μέλλον γι' αυτό το, νησί. Δηλαδή να αποτελέσει την πρώτη χωματερή για να απόβλητα στην Ευρώπη. Θέλω επισήμως να ζητήσω από την Κομισιόν να προσέξει και να παρέμβει πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λάμπρος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, η Ευρώπη βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις βίας. Θέλω να πιστεύω πως όλοι καταδικάζουμε τη βία και την τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται. Στην Ελλάδα δυστυχώς μόνο με λόγια και όχι με πράξεις. Από την ημέρα της εκλογής μας, οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή δεχόμαστε απειλητικά μηνύματα με επιστολή μας στον υπουργό προστασίας του πολίτη και στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας ενημερώσαμε για το γεγονός και ζητήσαμε μέτρα προστασίας τόσο για εμάς όσο και για τους τοπικούς βοηθούς που εργάζονται στα γραφεία μας. δυστυχώς δεν λάβαμε καμία απάντηση. καταγγέλλω ότι στις 24 δεκεμβρίου άγνωστοι έγραψαν με σπρέι απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής μας στους τοίχους και στην είσοδο των γραφείων μας. η αστυνομία απλώ κατέγραψε το συμβάν. στι 25 Δεκεμβρίου ξημερώματα Χριστουγέννων τη νύχτα άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο με αποτέλεσμα να υποστούν υλικέ ζημιέ στα γραφεία μα. Τόσο ο πολιτικό κόσμο τη χώρα όσο και τα μέσα μαζική ενημέρωση αποσιώπησαν το γεγονό. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στήριξή του για να πράξει όσο οφείλει η ελληνική κυβέρνηση και επιτέλους να τοποθετηθεί 24 ώρη φύλαξη στα γραφεία μας έτσι ώστε οι συνεργάτες μας και εμείς να μπορούμε απερίσπαστοι να ασχοληθούμε με το έργο μας. Ήδη ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή θρυνεί δύο θύματα από τρομοκρατική επίθεση την 1η Νοέμβρη 2013. Ελπίζω να μην θρυνήσουμε κι άλλα θύματα και μετά μπροστά στις κάμερες να λέμε «Είμαι κι εγώ Σαρλί». Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε εκλογές 25 Ιανουαρίου και αυτό δίνει την ευκαιρία σε διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωση να επαναφέρουν το θέμα του λεγόμενου Brexit, δηλαδή της αναγκαστικής εξόδου από την Ευρωζώνη. Μάλιστα, ορισμένοι διεθνεί οίκοι δίνουν και ποσοστά τη τάξη του 25%. Θεωρώ ότι αν όλοι είμαστε συνεπεί, Έλληνε και Ευρωπαίοι συνάδελφοι, προς τις υποχρεώσεις μας όλα θα πάνε καλά και απαντώ έτσι και στις ανησυχίες για την, σε ορισμένους που συνδέουν την, την, ε, τα προβλήματα της Ελλάδας με το ευρώ. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και δεύτερον, να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους, να πάει από τα 30 στα 50 χρόνια, να πέσουν τα τοκοχρεωλήσια και να μπορέσει έτσι να αναπτυχθεί η οικονομία. Εάν είμαστε αποτελεσματικοί και γρήγοροι, θα προλάβουμε τις, αρνητικέ ε, εξελίξει αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία και θα εκμηδενήσουμε τις πιθανότητες για το λεγόμενο Brexit. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέτσο και συγγνώμη που σας είπα ότι πρέπει να συντομεύετε, δεν υπολόγισα σωστά το χρόνο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντάνιελ Μπούντα, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Άρα επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ρόζα Φων Χόενστάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε όλοι την κατάσταση όπου σε κάποια κράτη-μέλη οι κυβερνήσεις ε, ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ άλλες χώρες επιστρέφουν τους, ε, τους μετανάστες. Και θα ήθελα να μιλήσω για την υπόθεση Μούρτμπεκ και Τεμπάγεφ που έλαβε το άσυλο στην Πολωνία και τώρα κινδυνεύει να επιστραφεί στην χώρα προέλευσή του από την Ισπανία. Θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους σας να μην ε, στέλνετε κόσμο που, που κινδυνεύει να βασανιστεί στη χώρα προέλευση του πίσω. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτοί που έχουν λάβει το άσυλο σε ένα από τα κράτη-μέλη να προστατεύονται σε ολόκληρη την Ένωση. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπούτα, θα έρθει η σειρά σας στον επόμενο γύρο. Ο κύριος ε, Τονίνα. Στην αρχή αυτού του χρόνου στην ε, Κροατία έπαψε να υπάρχει κατηγορία των ε, αλλιέων ε, μικρομεσαίου μεγέθους οι οποίοι στήριζαν την διαβίωσή τους σε μικρά λευτικά σκάφη ο στόχος ε, διατήρησης της ε, σταθερότητας των αλευτικών αποθεμάτων είναι αδιαφυσβήτητος. Ωστόσο, είναι... Ε, ωστόσο, γιατί θα πρέπει οι μικροί αλείς να θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτό το φαινόμενο. Η επίλυση είναι καλύτερος έλεγχος, όχι απαγόρευση η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει τα επαγγελματικά σκάφη. Αλλά υπάρχει και ένας, και ένας ο οποίος αναφέρει την ποικιλία των ελευτικών σκαφών ε, στο επίπεδο της μικρομεσαίας αλίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι ε, περνάει από το χέρι μας ώστε να διατηρήσουμε αυτή την αλία του μικρού και μεσαίου, ε, της μικρής και μεσαίας κλίμακας. Η κυρία Κέγκε. Ε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη που μίλησε στο Παρίσι θα πρέπει να είναι συνεπής και να αναλάβει μια έκτακτη ευθύνη όσον αφορά την υπεράσπιση της ελευθεροτυπίας της και ελεύθερης έκφρασης για να βοηθήσει όλες τις χώρες ε, ε, να αντιπαρέλθει ε, στις ακρότητες. Πριν από λίγες μέρες αποδόθηκε το βραβείο Σαχάροφ στον δόκτορα Μουγουέμπε και λίγες μέρες μετά πάγωσαν οι λογαριασμοί του νοσοκομείου το οποίο διευθύνει στο Κονγκό. Εμείς πρέπει να είμαστε υπέρ της της ε, παραβίασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως συμβαίνει τώρα στην, ε, δημοκρατική, στην λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Πρέπει να μιλάμε και για την Ιγυρία που έχει πέσει στα χέρια του Μπόκο Χαράμ και είμαι ευτυχή για την απόφαση που λήφθη σήμερα από το Κοινοβούλιο για να συνεχίσουμε με ψήφισμα σε αυτό το θέμα. Και άλλε επιθέσει και άλλοι θάνατοι. Αυτή τη στιγμή έγινε επίθεση εναντίον ενό χωριού στο Καμερούν. Δεν πρέπει να λείψει η ελπίδα την οποία ενσωμάτωσε πριν από λίγε μέρε ένα κοριτσάκι Μητσοτάκη, το οποίο ε, ε, ε, αρνήθηκε να πέσει θύμα της, της έκρηξης και αντιτέθηκε στις αρχές. Θα πρέπει η Ευρώπη να στείλει μια διεθνή task force στην Αφρική. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μάρκος Πρέτσελ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τον ε, σεβασμό μου στους ε, γελιογράφους ε, και λοιπούς ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν για την υπηρεσία που προσέφεραν στην κοινωνία μας και στους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον και στα υπόλοιπα θύματα που έπεσαν γιατί είναι μέλος της κοινωνίας που μισούν τόσο πολύ οι τρομοκράτες αυτοί. Συμπάσχω με τους συγγενείς των θυμάτων. Ανησυχώ όμως πως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ασχολείται με την επίρρηψη ευθυνών ενώ δεν υπάρχει κάποια ενότητα η οποία θα αντιταχθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά συζητάμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι που θα έχουμε. Για την διαφύλαξη κατόπιν αυτών των αξιών για να είναι ισχυρή η κοινωνία μας ε, κατά αυτών των ακραίων που μας απειλούν με τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αγγέλικα Μλίναρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι νιώθουμε μεγάλη ανησυχία και φόβο γιατί δεν ξέρουμε βεβαίως ε, τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε και έγινε σαφές πλέον πως η ελευθερία λόγου και η δημοκρατία είναι αξίες που πρέπει να υπερασπιστούμε και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνία ε, η οποία θα αξίζει πραγματικά να παλέψουμε για, αυτούν, γιατί, για αυτήν. Γιατί βεβαίως η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο. Η επαναφορά της θανατικής ποινής, η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και άλλα πράγματα που ακούγονται από δεξιά δεν είναι μόνο λανθασμένες απαντήσεις στην τρομοκρατία αλλά είναι και λαθασμένος τρόπος αντιμετώπισης. Χρειαζόμαστε περισσότερο κράτος δικαίου και δημοκρατία. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα πούμε. Ευχαριστώ, Ντανιέλ Μπούντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. η Ρουμανία συχνά όσον αφορά την ένταξη στην Σέγγεν αντιμετωπίζεται ως κράτος ε, δεύτερης ε, κατηγορίας. Ε, μας έλεγαν πως δεν πληρούνται οι απαιτήσει ασφαλής στα σύνορά μα. Κάτι το οποίο σήμερα συμβαίνει όμως και το αναγνωρίζουν όλοι. Η Ρουμανία ε, προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή και στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά η ένταξη στην Σέγγεν δεν γίνεται χωρίς καμία αιτιολογία. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο για μια Ευρώπη η οποία παίρνει στα σοβαρά τον ε, εαυτό της. Νομίζω έτσι επηρεάζεται και η μετακίνηση Ρουμάνων πολιτών και αγαθών Πρέπει να το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα. Η Ρουμανία θα πρέπει να έχει ίση μεταχείριση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο δικαίωμα της Ρουμανίας, αλλά και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μίλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το 2011 είχαμε την στρατηγική της ε, Ρώμης ε, πάρα πολλά έγγραφα αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει σήμερα στην Ευρώπη δεν έχει γίνει τίποτα για τους Ρωμά εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις και παρά το γεγονός ε, αυτό δεν θεωρώ πως η Κομισιόν ε, παίρνει τα πράγματα σοβαρά και δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνο για τα ζητήματα Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μιλάμε εμείς εδώ πέρα, ε, κυρία Πρόεδρε, εσείς και εγώ, ως Ευρωπαίοι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ζήτημα αυτό πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίτερ Μίλλερ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπέατριξ Φων Στόρχε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αυτοί που κάνουν την πολιτική. Ε, αρκεί ε, μία λέξη και μία τέτοια λέξη είναι η Grexit, το το οποίο εκφέρεται από ε, κύκλους της Γερμανίας ή τουλάχιστον δεν διαψεύδεται εκεί. Αλλά ε, χρησιμοποιείται η έννοια αυτή για να εξαπατηθούν οι Γερμανοί ψηφοφόροι οι οποίοι πρόκειται να ψηφίσουν για το τρίτο πακέτο αδειάση για την Ελλάδα και αυτός ο οποίος απειλείται είναι ο Έλληνας ψηφοφόρος ο οποίος δεν θα πρέπει να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για κατάφορη παρέμβαση στις δημοκρατικές εκλογές μιας δημοκρατικής χώρας και θεωρώ ότι αυτό είναι, υπόγεια, είναι μια υπόγεια μη δημοκρατική κίνηση. Ε, και πραγματικά δεν είναι ένα νόμισμα στην καρδιά της Ευρώπης αλλά η δημοκρατία αυτή η οποία διακυβεύεται εδώ και ας την προστατεύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σίλβιο Μπουζόη. Η Charlie Hebdo το περιοδικό Charlie Hebdo έπεσε θύμα μιας ε, τρομοκρατικής ε, επίθεσης και όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται κάτω από την κατάσταση σοκ. Η, πορεία χθε στο Παρίσι απέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν αφήνονται να αποδυναμωθούν από την ε, τρομοκρατία αλλά θέλουν να παλέψουν για την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε ε, κατά της ε, μυσαλλοδοξία και θα πρέπει να ενισχύσουμε τους οργανισμούς εκείνους που προσπαθούν να εξαλείψουν την τρομοκρατία και θα πρέπει να χαράξουμε στρατηγικέ για να παλύψουμε τα αίτια της τρομοκρατίας. Ε, θα ήθελα να εκφράσω θερμά μου ε, συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων. Je suis Charlie. Επόμενος ο μιλητής είναι ο κύριος ε, Μπαγιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. είχε δοθεί μία συνέντευξη η οποία αναφερόταν στο κίνδυνο του αποπληθαρισμού. Ε, και ε, έγινε λόγος για την αύξηση της ε, ανεργίας. Η πολιτική λιτότητας αποδεικνύει σήμερα την εμβέλεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της πολιτικής ε, λιτότητας. Ένα πρώτο βήμα ανάκαμψης έγινε μέσω του σχεδίου το οποίο προτείνει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να πάμε ε, πιο πέρα και θεωρώ ότι είναι ουσιώδες ε, να γίνουν επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να αλλάξει ο προϋπολογισμός του ελλείμματος και θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει το δικό της μερίδιο όσον αφορά ε, τον κίνδυνο του αποπληθαρισμού. Ε, ε, θα πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις και να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαγιέ. Η τελευταία ομιλήτρια στο κατάλογό μου είναι η κυρία Γκαρσία, Αγιλέρα Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταγγείλω την κατάσταση των θυμάτων του φρακισμού στην ε, Ισπανία η αναγνώριση ενός, εκ μέρους ενός λαού της ιστορικής του μοίρας ε, είναι δημοκρατική ευθύνη μιας χώρας η οδύνη των θυμάτων του φρακισμού ε, στην ε, Ισπανία ε, είναι τεράστια. Πολλά από αυτά τα θύματα, η σωρία αυτών των θυμάτων δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν γιατί βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους. Υπάρχει ένας νόμος που προβλέπει τέτοιου είδου ενέργειες αλλά ο οποίο έχει ε, εξοδερθεί από την ε, παρούσα κυβέρνηση της Ισπανίας ιδιαίτερα στην ε, περιοχή της Ανταλωσίας και επιτρέπει να μην υπάρξει κανένας χώρος για την αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά τα θύματα του φραγκισμού στην Ισπανία. Θα ήθελα λοιπόν να καταγγείλω αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μου, στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λίλερα Γαρσία. Ε, ολοκληρώνεται τώρα ο κύκλος των ομιλητών για τις παρεμβάσεις ενός ε, λεπτού. Η συνεδρίαση Ολομέλειας θα λάβει χώρα αύριο την ε, Τρίτη. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιοποιηθεί και βρίσκεται και στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση. καλό βράδυ.